Είναι σαφές ότι απαιτείται επικοινωνία ανάμεσα στα δύο μέρη. Είναι σαφές ότι το Ισραήλ είναι σημαντική χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τις διαφορές και να αποκαταστήσουμε την ειρήνη, να καταστήσουμε το Ισραήλ ασφαλές και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει σημαντική στην περιοχή και αντικειμενικός διαιτητής για τα προβλήματα της περιοχής, προωθώντας την μη βία, ε, τη δικαιοσύνη και τις προηγούμενες νομικές υποχρεώσεις, συμφωνίες και συνθήκες. Έτσι λοιπόν η λύση των δύο κρατών θα επιτρέψει στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη να ζήσουν μέσα σε σύνορα αναγνωρισμένα και ασφαλή. Να θυμίσω βέβαια ότι τα σώματα του Ισραήλ, ε, του, συγγνώμη, τα σώματα των ε, Ηνωμένων Εθνών έχουν καταφερθεί εναντίον του Ισραήλ ε, με πολλαπλό τρόπο στο παρελθόν. Δεν είναι αυτό σωστό. Έτσι και αλλιώς το Ισραήλ είναι η πραγματική δημοκρατία σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Ευχαριστούμε κυρία Μαρία Ρένα εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών. Σας ευχαριστώ πολύ. Η δημιουργία επικισμών ε, στις Παλαιστινιακές ε, περιοχές ε, και στην Ιερουσαλήμ δεν έχει καμία νομική βάση. Αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και σημαντικότατο εμπόδιο στην υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών για μια βιώσιμη ειρήνη. Είναι η παράγραφος 1 ε, του ψηφίσματο 2433 του Συμβουλίου Ασφαλεία, τα υψίπεδα του Γκολάν και ε, η Δυτική Όχθη συμπεριλαμβανομένη Ανατολική Ιερουσαλήμ δεν είναι κομμάτι του Ισραήλ. Ε, άρθρο 16 της σχετικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είναι αμέτρητες οι πηγές του δικαίου ευρωπαϊκού και διεθνούς που καταγγέλει την παρανομία των επικισμών. Έτσι λοιπόν η ανακοίνωση του κ. Πομπέου στις 18 Νοεμβρίου δεν είναι παρά μια πρόκληση επιπλέον. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε να τηρούμε το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και ευχαριστώ την κυρία Μογκερίνη για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει προς αυτές τις δύο κατευθύνσεις. Σεβασμός του διεθνούς δικαίου, σύνορα του 67 και σεβασμό του ευρωπαϊκού δικαίου. Το δικαστήριο μα υπενθύμησε στι 12 Νοεμβρίου υποχρεώνει τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να επισημαίνουν τα προϊόντα με ακρίβεια όταν προέρχονται από τα Ισραηλινά Παλαιστινιακά εδάφη και από του επικισμού. Εδώ είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εσεί είστε από την Επιτροπή. Πρέπει να σεβόμαστε το διεθνέ δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Είναι καθήκον μα και ευθύνη μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενο ομιλητή ο κύριο Νάρτ από το Ρινιού. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριος ε, στόχος των διεθνών σχέσεων δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πολιτική ισχύς. Το Ισραήλ συστηματικά παραβιάζει τα ψεφίσματα των ΗΕ, την Τέταρτη Σύμβαση της Γενέβης και την ίδια τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει κατά λέξη ότι βασίζεται στις δημοκρατικές αρχές και στα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελώντας ένα πολύ βασικό στοιχείο της συμφωνίας. Ρωτάω λοιπόν, πότε θα πετήσουμε την τήρηση της συμφωνίας αυτής. Ναι, συνεργασία, αλλά εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, μας αγνοεί και ο σύμμαχός μας, οι Ηνωμένε Πολιτείε αγνοούν το Όσλο και επιτρέπουν την κυριαρχία του Ισραήλ στα κατεχόμενα. Δεν είμαστε συνεπείς και δεν μας σέβονται και δεν μας σέβονται γιατί δεν σεβόμαστε εμείς οι ίδιοι τους αυτούς μας. 50 χρόνια κατοχής είναι κάτι απαράδεκτο. Οι καταδίκες τελικά δεν λειτουργούν, δεν βοηθάνε σε τίποτα. Να περάσουμε στις πράξεις. Ευχαριστούμε. Σατούρεκ, εκ μέρους των Πρασίνων τώρα. Ευχαριστώ. Είπατε εκπρόσωποι, τη στιγμή που οι Ηνωμένε Πολιτείε ξανασυντάσσουν το διεθνές δίκαιο, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα με αυτό, η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαναλαμβάνει τις ίδιες θέσεις. Δηλαδή, μιλάει για τους επικισμούς στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στον Κολάν, και η απόφαση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Γνωρίζουμε ότι ο επικισμός εμποδίζει την ειρήνη. Από το 1967 ξανά και ξανά από 16.000 έχουμε περάσει 460 έπικους. Αυτά είναι τα στοιχεία του 2018 της Peace Now που είναι του Ισραήλ η οργάνωση αυτή. Η Ευρώπη λοιπόν εμένει στις αρχές της. Ναι, αλλά έφτασε η στιγμή για την Ευρώπη μας να σταθεί στο ύψο τη και να συνεισφέρει συγκεκριμένα στην επίτευξη της ειρήνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι είναι υπέρ του δικαίου, τώρα πρέπει να το εφαρμόσει και να φροντίσει να τηρηθεί. Έχουμε τα μέσα να το κάνουμε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι θα υπάρξει σύμβαση των προϊόντων που έρχονται από τους επικισμούς και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχει το θάρρος να πάει ακόμα πιο μακριά και να φροντίσει να γίνεται σεβαστό το διεθνέ δίκαιο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λίτσι, μη εγγεγραμμένος. Έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Μογκερίνη. Όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επικισμοί του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη δεν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, όμως ε, το διεθνές δίκαιο επιβάλλει ε, ειδική ετικετοθεσία στα προϊόντα που προέρχονται από κατεχόμενα εδάφη. Γιατί ε, δεν κάνει το ίδιο η Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες 200 αμφισβητούμενες ε, περιοχές στον κόσμο. Οι Σουνίτες δεν διαμαρτυρήθηκαν έτσι και αλλιώς ιδιαίτερα για την Αμερικανική απόφαση και το βασικό τους πρόβλημα είναι το Ιράν ο εχθρός όλων είναι η τρομοκρατία. Ε, θέλουμε να αποφύγουμε φυσικά και ε, αντίστοιχες ενέργειες με την Τουρκία, την Ισλαμική Τουρκία που κατέχει την Κύπρο. Ευχαριστώ. Ο επόμενος, ο Βόντελ, για το ECR. Νομίζω ότι το θέμα αυτό, λέει ο κύριος Βόντρα, αφορά γενικά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Το Ισραήλ είναι βασικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τομέα της ασφάλειας και στον τομέα της οικονομίας. Έχουμε ανάγκη το Ισραήλ και το Ισραήλ έχει εμάς ανάγκη. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρηθεί το Ισραήλ, ε, να θεωρηθούμε και από το Ισραήλ ε, ως αντικειμενικός διαιτητής και δεν θα πρέπει να παρεξηγηθεί η θέση μας. Η ειρήνη ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη θα υπάρξει όταν αποκτήσουν μία ηγεσία και μία κυβέρνηση οι Παλαιστίνοι εναντίον της βίας και γι' αυτό η Ευρώπη δεν θα πρέπει να πληρώνει χρήματα αλλά θα πρέπει να επηρεάζει και ο μοχλός αυτός θα πρέπει να οδηγήσει στον τερματισμό ε, της συνεχούς ε, ενθάρρυνσης της Παλαιστινιακής ε, Αρχής όπως επίσης και να διακοπεί η ενίσχυση προς την Ούνρα η οποία με τη λειτουργία της ρίχνει λάδι στη φωτιά της σύγκρουσης. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Άντερσον από την ΚΟΕ. Συνάδελφοι, χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας σήμερα και παίρνω το λόγο στη συζήτηση αυτή. Πράγματι τα προϊόντα, η χημή και τα οροκυπευτικά που παράγονται στις κατηχόμενες περιοχές ε, θα πρέπει να τύχουν ειδική ε, ετικέτας, αλλά δεν αρκεί αυτή. Ε, θα πρέπει όλα τα προϊόντα τα οποία ενισχύονται ή μάλλον προέρχονται από περιοχές τις οποίες παράνομα κατέχει, ενισχύει οικονομικά και διατηρεί εν ζωή το Ισραήλ να μην μπορούν να εισάγονται το εμπόριο με τις παράνομες αυτές εγκαταστάσεις μας καθιστά συνενόχους του πολέμου εις βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Θα πρέπει να απαγορεύσουμε τις εισαγωγές και εν μέρη έχει γίνει αυτό, αλλά η Ιρλανδική κυβέρνηση δυστυχώς δεν βοηθά και συνεχίζει να εισάγει προϊόντα. Οι κυβερνήσεις της Ένωσης όπως και οι δικοί μου λέγουν ότι είναι υπέρ της λύσης των δύο κρατών αλλά παρόλα αυτά αποδέχονται την καταστροφική και επικίνδυνη πολιτική του Ισραήλ στον τομέα των επικισμών. Ακούμε συνεχώς για παραβιάσεις των δικαιωμάτων από πλευράς του Ισραήλ, αλλά παρόλα αυτά Δυστυχώς δεν βοηθάμε με τον τρόπο που πρέπει τους κατεχομένους, αλλά βοηθάμε αυτούς οι οποίοι τους κατέχουν. Συγγνώμη, δεν καταλάβετε καλά, είχατε ένα λεπτό. Επόμενος ομιλητής, ο συνάδελφος αντιπρόεδρος, ανεξαρτούς κ. Καστάλντο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Σε μια κίνηση αναμενόμενη μάλλον, ο Υπουργό Εξωτερικών Πομπέο ανακοίνωσε ριζική αλλαγή τη πολιτική των ΗΠΑ 18 Νοεμβρίου όσον αφορά του επικισμού στη Δυτική Όχθη, επιβεβαιώνοντα ότι δεν θα θεωρεί πλέον ότι είναι παράνομη ε, βάσει του διεθνού δικαίου. Με αυτή την ε, ε, απόφαση η διοίκηση των ΗΠΑ έπαψε να είναι αξιόπιστος διαμεσολαβητής ε, στην ε, διαφωνία αυτή στη Μέση Ανατολή και δεν συμμετέχει πλέον στη λύση των δύο ετών. Είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά εγώ θα ήθελα να είμαι επικοδομητικός με τη ΣΥΠΑ που παρετήθηκαν ουσιαστικά από το ρόλο τους τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ένα βήμα μπροστά, να αναγεννήσει από τις τάχτες μια διαδικασία ερηνευτική περίπλοκη αλλά αναγκαία ενώ ολόκληρη η Μέση Ανατολή φλέγεται, έχει μπει σε δεύτερο ε, ε προτεραιότητα η σύγκρουση Παλαιστινίων-Ισραήλ σαν να είναι κάτι που δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Αυτό είναι λάθος, ενώ είναι η βασικότερη ε, διαφορά ε, που υπάρχει και απαραίτητη συνθήκη για τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ύπατη εκπρόσωπο για το έργο τη και θα ήθελα να ζητήσω από τη νέα είπατε και τη νέα Κομισιόν να συνεχίσουν τι προσπάθειε με ε, νέες προτάσεις, ε, ρεαλιστικέ, νέε ελπίδες με σεβασμό του διεθνού δικαίου και των αποφάσεων του δικού μα δικαστηρίου και με συνοχή. Το, ε, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό για να υποστηρίξουμε τι αξίε μα. Αλλιώ θα χάσουμε άλλη μια ευκαιρία για την περιοχή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο ομιλητή, είναι ο κύριος Μάντλ. Εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει μία πολιτική, μία ηθική πτυχή, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά η συνολική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ηθική πτυχή κατά την απόψή μου είναι ότι μιλάμε για το μοναδικό Εβραϊκό κράτος στον πλανήτη, μιλάμε για το αρχαίο ε, για την αρχαία κατοικία των ε, Εβραίων όχι μόνο για δεκαετίες και αιώνες αλλά για χιλιάδες χρόνια. Ποιοι είμαστε εμείς λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα πάμε να κρίνουμε οποιονδήποτε Εβραίο που πάει να μείνει εκεί. Και μετά υπάρχει η πολιτική πτυχή. Αν απομονώσουμε το ζήτημα των επικισμών από όλα τα υπόλοιπα, αυτό σημαίνει ότι παραβιάζουμε την ειρηνευτική διαδικασία. Όχι ότι την υποστηρίζουμε, διότι δεν βλέπουμε παρά μία πτυχή από πολλές ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία πρέπει να είναι ε, αυτή ενό ειλικρινούς διαμεσολαβητή. Μιας δύναμης που υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια είναι αυτό το οποίο χρειάζεται το Ισραήλ και ότι η ασφάλεια είναι αυτό το οποίο απαιτείται. Γι' αυτό είναι σημαντικό το Ισραήλ να παραμείνει ε, στον έλεγχο των περιοχών αυτών που, από τις οποίες προέρχονται απειλές ε, για τον μη στρατιωτικό πληθυσμό του Ισραήλ και εφόσον υπάρχει ασφάλεια σε αυτές τις περιοχές αυτός ο έλεγχος Πρέπει να παραμείνει για να υπάρχει αυτή η ασφάλεια και η ειρηνευτική διαδικασία θα πρέπει να βοηθηθεί ω διαμεσολαβητή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο από ποτέ πρέπει να είναι να σταθεί στο πλευρό του Ισραήλ και να το υποστηρίζει. Είναι η μόνη δημοκρατία, το μόνο κράτο δικαίου στη Μέση Ανατολή. Κυρία Μογκερίνη, σα ευχαριστούμε για το έργο σας. Και εγώ θα ζητήσω αυτή η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπογραμμίζεται σαφώς και από το έργο σας και από τους διαδόχους σας. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Ινσύρ, εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε έχουμε δύο δημοκρατικές χώρες, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, που ειρηνικά να ζουν η μία δίπλα στην άλλη. Αυτό είναι ο στόχος μας. Αλλά για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να δέχονται και οι δύο πλευρές το διεθνές δίκαιο και κοινέ προδιαγραφές. Η κατάσταση που έχουμε σήμερα δεν είναι αυτό. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι διεθνεί παράγοντε όπω είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε που οδηγούν σε πόλωση αντί να προσπαθούν να βρουν μια λύση ε, μετακομίζοντα α πούμε την πρεσβεία του στην, ε, στα Ιεροσόλυμα ή με τι ε, δηλώσει που κάνουν που λένε ότι οι επικισμοί δεν είναι παράνομοι. Για να υπάρξουν δύο κράτη πρέπει να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη. Από το 2014 το προσπαθούμε και θα έπρεπε πολύ περισσότερες χώρες να το κάνουν. Ως αντιπρόεδρος για την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη, θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα. Πρόκειται για τα κατεχόμενα, πρόκειται για τους επικισμούς, αλλά πρόκειται και για τα προϊόντα της περιοχής. Πρόκειται επίσης για την ανθρωπιστική βοήθεια. Από το 2014 έχουμε υποδομές που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τις χώρες μέλη και καταστρέφονται από τον στρατό του Ισραήλ. Είναι απαράδεκτο αυτό, οπότε είναι απλό το ζήτημα. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην συμβαίνει αυτό και για να μην συνεχίζεται. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι θα υπάρξει κάποια αποζημίωση για όλα αυτά. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής, Κροσέλ, από τη Ρινιού. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για το ζήτημα της ε, πλαεστινής. Ε, ε, απομακρύνεται η λύση λόγω της απόφασης του κυρίου Τραμπ για την Ιερουσαλήμ και την κατάσταση των Ισραηλινών επικισμών. Η ανθρωπιστική κρίση εντείνεται. Η διεθνής κοινότητα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν δείχνει να έχει κάποιο ενδιαφέρον για μια βιώσιμη λύση και το status quo συνεχίζεται τους ε, κάνει μια χαρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να επιμείνει στη λύση των δύο κρατών και να ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει τους επικισμούς ε, στις ε, Παλαιστινιακές περιοχές. Να το απαιτήσει αυτό και να επιβάλλει να επανέλθουν όλοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια βιώσιμη λύση. Ανεξάρτητα από τις τελευταίες εξελίξεις, το ζήτημα αυτό δεν είναι δυνατόν να επιληθεί παρά μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Ντάουντινγκ από τους Πρασίνους. Αγαπητοί συναδελφοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επιτέλους να αποτελέσει τον βασικό διαμεσολαβητή μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Αυτό απαιτεί δέσμευση με το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι πολύ σημαντική. Τα προϊόντα από του παρανόμου επικισμού πρέπει να φέρουν τη σχετική επισήμανση πλέον και πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα βήματα για να υλοποιηθεί η απόφαση του δικαστηρίου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απαγορεύσει όλες τις εισαγωγές προϊόντων από τις επικισμένες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόμοια μέτρα έχουν ληφθεί για προϊόντα από την Κρυμαία, από τη Βορειοκύπρο, γιατί όχι από τους επικισμούς τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει επιγοντό να ε, δημοσιεύσουν ε, τη βάση δεδομένων με τις επιχειρήσεις ε, που λειτουργούν στους επικισμένες περιοχές και που κερδοσκοπούν από αυτή την ανάπτυξη. Οποιαδήποτε προσπάθεια νομιμοποίηση τη προσάρτηση αυτών των περιοχών και παραβίαση του διεθνού δικαίου θα πρέπει να έχει συγκεκριμένε συνέπειε. Και τέλο, θα ήθελα να ζητήσω από την ύπατη εκπρόσωπο και από τον διαδοχό τη να λάβουν και άλλα βήματα. Να μας πείτε τι άλλα βήματα μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε το διεθνές δίκαιο να αποτελεί το σημείο αναφοράς στην ειρνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ζαχραντήλ, εκ μέρους του ΙΣΕΑΡ. Εμείς όταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκινήσαμε να συζητάμε το θέμα του Ισραήλ, η κατάσταση έχει περιπλακεί ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει να κρατάμε μια ισορροπία, να δούμε τι είναι σημαντικό για την Ευρώπη και τι μπορεί να ε, δημιουργήσει πλέον εκτίματα στους Ευρωπαίους πολίτες αναγνωρίζοντας ότι το Ισραήλ είναι ίσως ο πιο σημαντικός περιφερειακός εταίρος, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφαλείας. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ εν πωλής είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, είναι ένα κράτος δικαίου, αν και δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ας δείξουμε λοιπόν την απαιτούμενη αλληλεγγύη προς το Ισραήλ, ιδιαίτερα στα πλαίσια της αυξανόμενης αντισημιτικής δραστηριότητας σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει ε, πιο ισόρροπα, δείχνοντας περισσότερη αλληλεγγύη ε, προς το Ισραήλ. Κρέσπο. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι συνένοχος του απαρτχάι της βάρος της Παλαιστίνης. Οι θεσμικές σχέσεις με υπηρεσίες του Ισραήλ που εμπλέκονται ε, στην καταστολή και την καταπίεση των Παλαιστινίων ε, μας καθιστά συνενόχους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σεβαστεί και τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα η οποία περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Συνεργασίας της με το Ισραήλ και να ακούσει, να η Ευρωπαϊκή Ένωση τα εγκλήματα εις βάρος των Παλαιστινίων και ε, μόνο η κοινωνία των πολιτών θέτει ξεκάθαρα τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευράς ε, ε, του Ισραήλ θα πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο κορυφής ε, για να τερματιστεί η καταστολή εις βάρος των Παλαιστινίων, να απαγορευτεί η εξαγωγή όπλων προς το Ισραήλ και να απαγορευθούν και οι εισαγωγές προϊόντων από τις παράνομα κατεχόμενες περιοχές. Ο κύριος Αλαβάνος, Νικολάου Αλαβάνος, 1,5 λεπτό. Η αναγνώριση από τις ΗΠΑ Αμερικής των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, η λεγόμενη Συμφωνία του αιώνα, που ουσιαστικά νομιμοποιεί την παράνομη απόσπαση και κατοχή Παλαιστινιακής γης από το Ισραήλ, η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα του Ισραήλ πρημοδοτούν την κλιμάκωση της επιθετικότητας απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό που υποφέρει δολοφονίες ακόμα και ανήλικων παιδιών επιθέσεις επικισμούς το τείχος του έσχους χιλιάδες πολιτικούς κρατουμένους. η ευρωπαϊκή ένωση έχει μεγάλες ευθύνες. κρατά ίσες αποστάσεις ταυτίζοντας το θύμα τον παλαιστινιακό λαό με το θήτη το ισραήλ. η στάση της δίνει άλοθη και τροφοδοτεί τη συνέχιση των θηριωδιών του ισραηλινού κράτους σε λωρίδα της γάζας και στη δυτική όχθη οι ελληνικές κυβερνήσεις της νέας δημοκρατίας και του σύριζα επίσης έχουν βαριές ευθύνες. επέκτηναν και αναβαθμίζουν συνεχώς την πολιτική οικονομική στρατιωτική συνεργασία με το ισραηλινό κράτος. υποστηρίζουμε το δίκαιο αγώνα του παλαιστινιακού λαού και απαιτούμε τη δημιουργία ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την ανατολική ιερουσαλήμ την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τα κατεχόμενα εδάφη την πάυση της επικιστικής δραστηριότητας και την αποχώρηση όλων των επίκων το γκρέμισμα του τείχους της ντροπής την επιστροφή των παλαιστινίων προσφύγων στις αιστείες τους την άμεση απελευθέρωση όλων των παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων να τεθούν τώρα σε ισχύ οι αποφάσεις των κοινοβουλίων 14 κρατών μελών ανάμεσά τους και η ελλάδα από το 2015 που έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος. This concludes the list of speakers for political groups. Uh, the blue card request can be... Υπάρχει μπλε κάρτα, όχι. Η κυρία Ασημακοπούλου τώρα έχει το λόγο. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Thank you, Mr. President. Madam High Representative, in this house I'm in a state... Ευχαριστώ. Σε αυτό τον οίκο έχω να πω ότι δεν είμαστε ούτε τυφλοί, ούτε κουφοί, ούτε ε, Μουγκή, ακούσαμε την θέση των ΗΠΑ, ε, το ακούσαμε από την την εκπρόσωπο όπως έχουμε ακούσει και στο παρελθόν και την περασμένη εβδομάδα και σίγουρα έχουμε ακούσει και τον πρόεδρο ε, Τραμπ και τον Υπουργό Εξωτερικών να μιλά πολύ σαφώς για το Ισραήλ. Δεν είμαστε τυφλοί. Εδώ και δεκαετίες βλέπουμε ματιρές επιθέσεις κατά Ισραηλινών πολιτών. Το έχω δει με τα δικά μου μάτια στο κιμπούτσι του Ναχάλα που είναι πολύ κοντά στην ε, ε, Γάζα όπου ο τετράχρονος Ντάνιελ σκοτώθηκε μες στο σπίτι του από ε, πυράβλους της Χαμάς. Το είδα με τα μάτια μου σε Ισραηλινά χωριά κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν όπου ο τοπικός πληθυσμός συχνά χρησιμοποιείται ως ανθρώπινη ασπίδα κατά των πυράβλων της Χεσμπολάχ ε, που χρησιμοποιούνται για επίθεση κατά Λαϊνών πολιτών. Είναι σαφές, το Ισραήλ έχει νόμιμα ε, ε, ανησυχίες για την ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει πολύ καθαρά στο παρελθόν ότι θέλει να προωθήσει τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή του Ισραήλ. Είναι ένας από τους στενότερους συμμάχους της Ευρώπης. Έχουμε κοινέ αξίες, κοινά συμφέροντα. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε τώρα είναι να προχωρήσουμε, να προωθήσουμε μια κοινή διμερή ατζέντα για να εμβαθύνουμε τους δεσμούς μας και είναι σαφές ότι ε, αυτό αποτελεί προτεραιότητα της νεοεκλεγής σας Επιτροπής. Η στενότερη συνεργασία θα μας βοηθήσει να προωθήσουμε την ειρήνη και θα βοηθήσει και την Ευρώπη να ενισχύσει το ρόλο της ως ειλικρινούς αξιοπρε... αξιο... αξιόπιστου δημοσιολαβήτη για την ειρήνη. Δεδομένη τη κατάσταση στο Ισραήλ, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να απέχει από το να παρεμβαίνει σε εσωτερικέ ε, πολιτικέ. Δεν είμαστε ούτε κουφοί ούτε ε, τυφλοί, αλλά μερικέ φορέ η ε, σιωπή είναι χρυσό. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε εδώ και καιρό βέβαια ο κατάλογο των ομιλητών εκ μέρου των πολιτικών ομάδων. Συγγνώμη, άλλαξε η Προεδρία και γι' αυτό μπερδεύτηκα. Ε, Αβραμ τώρα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Η κυρία Αβραμ. Καλωσορίζω την ισορροπημένη παρουσίαση της κυρίας Μογκερίνη για την κατάσταση στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη και θέλω να υπενθυμίσω στο σώμα και στο κόσμο που παρακολουθεί τη συζήτησή μας ότι το Ισραήλ είναι η μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή και ίσως θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες για να πείσουμε και άλλες χώρες στην περιοχή να ακολουθήσουν τον δρόμο της πραγματικής δημοκρατίας. Νομίζω ότι πολλά πράγματα θα ήταν πιο εύκολο να λυθούν στη Μέση Ανατολή και το θέμα της ειρήνης. Τώρα όσον αφορά τους επικισμούς. Πιστεύω ότι πρέπει να αποτελεί μέρο του πλαισίου διαπραγματεύσεων ανάμεσα στι Παλαιστινιακέ Αρχέ και τι Αρχέ του Ισραήλ. Το να στηρίζει κανεί τη μία πλευρά ποτέ δεν έχει βοηθήσει στην πρόθεση τη ειρήνη. Το Ισραήλ αποτελεί σύμμαχο, φίλο και εμπορικό εταίρο. Και όσον αφορά την ασφάλεια, η καινοτομία, η γεωργία, η καταπολέμηση τη τρομοκρατία ή ακόμη και η καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή είναι πράγματα ε, από τα οποία μόνο να υποφεληθούμε έχουμε από το Ισραήλ. Οπότε δεν είναι δυνατόν κάθε φορά να τα βάζουμε του φίλου μα, χωρί όμω, να πηγαίνουμε περισσότερο σε βάθο για το τι συμβαίνει στην περιοχή και χωρί να προσπαθούμε να κατανοήσουμε την πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να παραμείνει ένα να και ειλικρινή και μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε μια μακροχρόνια συμφωνία και ελπίζω και ειρήνη στην περιοχή. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Χόρουτ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συζητάμε αυτό το θέμα λίγες μέρες ε, μετά από ε, τη στιγμή που μαζί με τις ε, κυβερνήσεις της Αιγύπτου και Αλωνών αποφάσισε να απαγορεύσει το το Eurowatch. Οι καταστροφές είναι τεράστιες έτσι. Ο κύριος Παμπέο έκανε τις γνωστές δηλώσεις ότι επικισμοί στη δυτική όχθη δηλαδή δεν είναι απαραίτητα κάτι που στο διεθνές δίκαιο. Δεν είναι σωστό και έπειτα το ότι αλλάζουν την κατάσταση επιτόπου μειώνει τις πιθανότητες για τη λύση των δύο κρατών. Εδώ και καιρό έχουμε καταλήξει ότι είναι το μόνο σχέδιο που μπορεί να οδηγήσει στην ειρήνη ε, τα δύο κράτη. Φυσικά και έχει δικαίωμα το Ισραήλ να υπάρχει ως κράτος, αλλά το ίδιο δικαίωμα έχει και η Παλαιστίνη. Τηρεί τα κριτήρια του Μοντεβιδέο για να αποτελεί ανεξάρτητο κράτος εδώ και χρόνια και υπάρχουν και μετροπεθείς ηγέτες στην Δυτική Όχθη. Ελπίζω ε, κάποια στιγμή να το αναγνωρίσουμε αυτό και ότι αν υποστηρίξουμε αυτούς τους μετροπεθείς ηγέτες είναι το καλύτερο δώρο που έχουμε να κάνουμε και στο Ισραήλ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε αυτόν ακριβώς το δρόμο. Μάτζιτ, ένα λεπτό παρακαλώ. μου φίλοι. Το μήνυμά μου προς τους Παλαιστινίους οι οποίοι απειλούνται να εξαφανιστούν και να μην έχουν το δικαίωμα να υπάρχουν είναι το εξής. Υπάρχουν χιλιάδες Ευρωπαίοι οι οποίοι μεγάλωσαν υποκατοχή πίσω από σιδρά παραπετάσματα. Δεν σταματάει η καταστολή, ο εφιάλτης, τα βασανιστήρια. Οι Ευρωπαίοι αυτοί και οι σύμμαχοί τους, πολλοί ε, μπορεί να είναι αριστερή. Πάντω καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό και στηρίζω τον αγώνα σας. Και στους φίλους στο Κοινοβούλιο έχω να πω, δώστε στους Παλαιστινίους αυτό το οποίο θέλετε να έχετε κι εσείς. Η υπόσχεση πρέπει να είναι ότι δεν θέλετε κανένας να σκοτώνει τα παιδιά σας. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και εκεί. Αν είναι παράνομοι οι επικισμοί και τα προϊόντα τους, τότε αυτοί που προωθούν αυτά τα προϊόντα είναι εγκληματίες. Πρέπει να δράσουμε. Γι' αυτό μην ξεχνάμε και επαναλαμβάνω ότι είπε ο Νέλσον Μαντέλα που είπε ότι αν δεν έχουν ελευθερία οι Παλαιστίνοι, τότε δικιά μας η ελευθερία δεν είναι τέλεια, παραμένει ατελής. Ευχαριστώ. Η κυρία Μιχέλ, σε ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Μογκερίνη, προφανώς συμφωνούμε όλοι ότι η νομιμοποίηση της πολιτικής επικισμού του Νεδανιάχου από τον Πομπέο και τον Τραμπ ε, παραβιάζει το διεθνώς ε, δίκαιο. Οι ε, εκτοπισμοί πληθυσμών θα είναι ο επόμενος γύρος. Έχουμε ένα νέο κύμα αναγνώρισης της Παλαιστίνης με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι ο νέος στόχος ε, της ε, πολιτικής ε, για Μέση Ανατολή. Αυτή η διαδικασία ειρήνης που αποτυγχάνει διαρκώς θα πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί με μια ειρηνευτική λύση για τη Συρία για όλη την περιοχή. Πόσο αξιόπιστη είναι η διπλωματία μας στη Μέση Ανατολή όταν από την άλλη πλευρά χρησιμοποιούμε μια πολιτική αποκλεισμού προς την Τουρκία και τη Λιβύη. Δεν είμαστε αξιόπιστοι όταν τα κράτη-μέλη παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο με εξαγωγές όπλων και εκπαίδευση δυναμεών ασφαλείας. Χρειαζόμαστε μια διεθνή ειρηνευτική διάσκεψη για να δώσουμε πραγματικές απαντήσεις. One Ένα λεπτό, ο κύριος Μίξερ. Είπατε εκπρόσωπε αγαπητή Φεντερίκα, ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική σας συνεργασία την τελευταία αιτία και για την προσωπική σας δέσμευση να βρείτε μια δίκαιη βιώσιμη λύση σε αυτή την αιώνια διαμάχη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων και ευχαριστούμε για τη δέσμευσή σα ε, να διατηρήσετε την ενότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη δική μα προσέγγιση σε αυτή την ειρηνευτική διαδικασία. Η διαπραγμάτευση μια λύση δύο κρατών είναι ο μόνο τρόπο να επιληθεί η διαμάχη και ο η ε, πιστική λύση που μπορεί να καθησυχάσει ε, τις ανησυχίες ασφαλείας του Ισραήλ που δικαίως έχει και τις ε, ανησυχίες ε, της Παλαιστίνης για ένα κράτος. Η διαπραγμάτευση αυτή ε, ε, ε, υπήρξε, διακρίθηκε από συνοχή μέχρι σήμερα και πρέπει να παραμείνει έτσι. Ο επικισμό αποτελεί εμπόδιο στην ειρηνευτική διαδικασία. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σαφέστατοι στη θέση μα όσον αφορά αυτέ τι δράσει. Το ίδιο ισχύει και για την ενθάρρυνση τέτοιων δραστηριοτήτων από τι πρόσφατε δηλώσει των ΗΠΑ όσον αφορά του επικισμού. Δεν πιστεύω ότι μονομερεί δράσει που σαφώ δεν συνάδουν με το διεθνέ δίκαιο ε, συμφέρουν κανέναν από άποψη ασφάλειας ε, μακροχρόνια. Ευχαριστώ ο κύριος Μπάουσα Ένα λεπτό. Νομίζω ότι η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου είναι υποχρέωση όλων των κρατών και δεν μπορεί το Ισραήλ να είναι μια εξαίρεση. Με ανησυχεί ε, αυτή τη στιγμή η συμπεριφορά των ε, πλευρών ε, που εμπλέκονται στην διαφορά και πώς αντιδρούν στα θέματα τα οποία μπορεί να δημιουργεί το Ισραήλ. Η άνοδος του αντισημιτισμού σαν παράδειγμα είναι κάτι το ανησυχητικό. υπάρχουν διακρίσεις και προβλήματα για συγκεκριμένες θρησκευτικέ κοινότητες σε ένα μεγάλο ποσοστό των πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε ακριβώς και το τι δημιουργήθηκε σε μια, το πρόβλημα που εμφανίστηκε στη γερμανική πόλη του Χάλε ε, στα πλαίσια της εορτής ε, ε, το Ιόμ Κιπούρ. Είναι σαφές ότι οι, οι Ισραηλίτες δεν αισθάνονται ασφαλείς στην χώρα τους και γι' αυτό ακριβώς απαιτείται περαιτέρω επέμβαση και βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση των ηπα προσπαθεί να νομιμοποιήσει τις απαράδεκτες πολιτικές του ισραήλ. προκλητικά χαρακτηρίζει ως νόμιμους τους ισραηλινούς επικισμούς στην κατοχόμενη παλαιστίνη ενώ προηγουμένως μεταφέρει την πρεσβεία της στην ιερουσαλήμ και αναγνώρισε την κυριαρχία του ισραήλ στα υψώματα κολάν. την ίδια ώρα το ισραήλ επεκτείνει διαρκώς τους επικισμούς οι επικυκλιζανές δυνάμεις ασφάλειας συνεχίζουν τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων των παλαιστινίων. η ευρωπαϊκή ένωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι απαθής. πρέπει να ασκήσει πιέσει στο ισραήλ προκειμένου να τερματίσει την πολιτική των επικισμών και να δεσμευτεί σε ένα οδικό χάρτη για την ειρήνη και λύση εις τη βάση δύο κρατών. από το βήμα αυτό καλώ και την κυβέρνηση της χώρας μου της κυπριακής δημοκρατίας να καταγγέλνει τις ενέργειες των ηπα και του ισραήλ. ο οπικισμός συνιστά έγκλημα πολέμου. Κύριε Σάντος, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ε, κυρία είπατε εκπρόσωπε, κύριε Πρόεδρε. Σε αυτή την τελική σας ε, ημέρα εδώ στο Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια μας. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τα ακόλουθα λόγια που πρόσφατα δημοσιεύτηκαν για να πούμε τα πράγματα με απλό και άμεσο τρόπο. Η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί αφενός η ελευθερία για τους Παλαιστινίους, αυτοδιάθεση και ανάπτυξη αφετέρου το δικαίωμα των Ισραηλινών ε, για ειρήνη και ασφάλεια οποιαδήποτε θέση ενάντια σε αυτή όπως βλέπουμε όταν οι ΙΠΑ για παράδειγμα νομιμοποιούν επικισμούς ε, σαν ήταν νόμιμοι και όταν μετακινούν, ε, μεταφέρουν την ε, πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ αντίκειται του διεθνούς δικαίου και υπονομεύει την επίλυση της Ισραηλο-Παλαιστινιακής διαμάχης. και υπονομεύει οποιαδήποτε ιδέα ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πάει πιο πέρα από τα λόγια και να αρχίσει να δρά να, για να βρεθούν τρόποι να υλοποιηθεί η Συμφωνία του Όσλο, όπω και το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του 2016. Ευχαριστούμε ο κύριος Φίλομσεν. Ένα λεπτό. Πραγματι η στάση του Ισραήλ στα Παλαιστινιακά εδάφη είναι μια στάση που παραβιάζει ξεκάθαρα το διεθνές δίκαιο. Και δεν είναι απλώς αυτό. Στην ουσία είναι ένας τρόπος δημιουργίας περαιτέρω εμποδίων στις ειρηνευτικές διαδικασίες. Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου ε, στην ουσία παραβιάζουν συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει την πλήρη απαγόρευση προϊόντων που προέρχονται από τα κατεχόμενα εδάφη. Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους είναι κάτι το θεμελιώδες. Πρέπει να ζητήσουμε από τους Παλαιστινίους να ζήσουν πια ελεύθεροι. Ο κύριος Σαντσέζα Νομίζω ότι έχει ξεφύγει πλέον η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και ε, στην ουσία καλύπτουν νομικά με, συγκεκριμένες, ε, με συγκεκριμένα επιχειρήματα ε, εδάφη τα οποία είχαν κάποτε ρυθμιστεί με τις συμφωνίες του Ελσίνκη. θα μπορούσαμε να δεχθούμε ότι η Τουρκία σε λίγα χρόνια θα μπορούσε να είναι κάτοχος των περιοχών τις οποίες ελέγχει σήμερα νόμιμα. Το ίδιο συμβαίνει σήμερα με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Εμείς δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να μετατρέψουμε ακριβώς το αποτέλεσμα μιας βίαιης σύγκρουσης σε νόμιμη κατοχή είναι λοιπόν όχι μια απλή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, είναι μια κατά μέτωπον επίθεση πολιτική αυτή στον ανθρώπινο πολιτισμό. Ο κύριος Μαγιορίνο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Φεντερίκα για όλα εσύ κάνει μέχρι τώρα. Με πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία βλέπουμε την κατάσταση που διαμορφώνεται εδώ και καιρό στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη επιβάλλεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα να αντιδράσει ξεκάθαρα έτσι ώστε να ανακτήσουμε την πορεία που θα οδηγήσει στη λογική των δύο λαών, δύο κρατών. Είναι απαραίτητο χωρίς αυτό να μας κάνει να αποκλίνουμε από τις απόψεις μας. Θα πρέπει να υπάρξει αμοιβαίος σεβασμός και αμοιβαίος σεβασμός και του δικαιώματος του Ισραήλ να ζήσει εν ασφαλεία σε διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα και ακριβώς το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τον Παλαιστινιακό λαό, τον οποίον τα όρια θα πρέπει να αναγνωριστούν στα πλαίσια της αναγνώρισης του κράτους τους, της κυριαρχίας τους, της νομιμότητάς τους και οτιδήποτε είναι ενάντια με αυτά είναι απαράδεκτο. Η πολιτική Νετανιάχου για τους επικισμούς είναι κάτι το απόλυτα αποσταθεροποιητικό. Είναι πραγματικά μια αδικαιολόγητη μορφή πίεσης αντίθετη με το διεθνές δίκαιο. Η κυρία Φαγιόν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώνει σιγά σιγά η θητεία σας και ευχαριστούμε για την εξαιρετική δουλειά, αγαπητή Φεντερίκα. Η συζήτηση για την κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη δυστυχώς ε, χαρακτηρίζεται από βία. Πάνω από 39 θύματα είχαν οι επιθέσει του Ισραήλ στη Γάζα το βλέπουμε διαρκώ. Και η λύση βρίσκεται στο διάλογο και στην ειρηνευτική διαδικασία, αλλά μέχρι στιγμή δεν έχει επιτύχει. Έχει δηλητηριαστεί, παρεμποδίζεται από τα μονομερή ε, μέτρα των ΗΠΑ και του Πρόεδρου Τραμπ ε, για τη θέση που έχει λάβει όσον αφορά τους παρανόμους επικισμούς ε, στη Δυτική Όχθη. Αυτό παρεμποδίζει το να δοθεί μια απάντηση. Έχουμε και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αναφέρει ότι πρέπει να επισημένονται τα προϊόντα από τους παρανόμους επικισμούς. Είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου, είναι έγκλημα πολέμου ε, ο επικισμός αυτός και τα προϊόντα που παράγονται εκεί είναι παράνομα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν έχουν θέση στην Ευρώπη. Η Κομισιόν θα πρέπει αμέσως να δράσει ούτως ώστε να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση του δικαστήριου ώστε το Ισραήλ ε, να μην έχει τέτοιο δικαίωμα και να ή μην υπονομεύει την ειρηνευτική λύση. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Αντιπρόεδρε, θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την πολιτική ε κυρια Διπρόεδρε, ήταν σαφής πάντα μέχρι τώρα και ελπίζω να παραμείνει έτσι. Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να υπονομεύσει το διεθνές δίκαιο αποτελεί μια πραγματική απειλή στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Αντί να ενώσουμε δυνάμεις για να βρεθεί μια ειρηνική λύση για δύο κράτη, η κατάσταση επιδεινώνεται και απειλείται η ήδη έφραστη κατάσταση όσον αφορά την προοπτική των δύο κρατών δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου. Γι' αυτό πρέπει να σταματήσουν όλες οι δραστηριότητε που έχουν να κάνουν με τους επικισμούς, να απαγορευτούν επίσης τα προϊόντα που προέρχονται από τους επικισμούς και φτάνουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Αλλιώς είναι σαν να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Η βία επίσης πρέπει να σταματήσει. Ο κόσμος πρέπει να νιώθει ασφαλής και να προστατεύεται και η κλιμάκωση να αποφευθεί πάση θυσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τώρα με τη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Ο κύριος Κάλαχαν έχει πρώτο το λόγο. Θέλω να πω ευθύ εξ αρχή ότι σέβομαι το δικαίωμα του Ισραήλ να προστατεύει τον εαυτό του, να υπάρχει και να ζει σε ειρήνη. Όμω επισκέφθηκα τη Δυτική όχθη και είδα τι σημαίνει κατοχή από πρώτο χέρι. Υπονομεύει την ίδια την ύπαρξη του Παλαιστινιακού κράτους. Μην έχουμε ψευδεστήσεις. Η ιδέα ότι το Ισραήλ μπορεί να συνεχίσει να χτίζει στα Παλαιστινιακά εδάφη υπονομεύει οποιαδήποτε πιθανότητα για ειρηνική λύση. Το Παλαιστινιακό κράτος διαλύεται σιγά σιγά μπροστά στα μάτια μας. Και ο απεσταλμένος του Ηνωμένων Εθνών δεν μιλάει με τους Παλαιστινίους. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει έναν πιο ενεργό ρόλο. Ναι, έχει δικαίωμα το Ισραήλ να υπάρχει, αλλά συγχρόνω πρέπει να διασφαλίσουμε, να διασφαλίσουμε ότι η λύση των δύο κρατών αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθα για οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία. Στο Ελλαδικό Κοινοβούλιο το είχα πει πριν από χρόνια όσον αφορά τους παρανομούς επικισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να το κοιτάξει. Και όχι μόνο στην Δυτική Όχθη, αλλά παντού όπου αυτοί υπάρχουν ανά τον κόσμο. Ευχαριστούμε. Ριτζίνσκι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Κύρια, είπατε εκπρόσωπε, το 1492 όταν εκδιώχθηκαν από την Ισπανία και την Πορτογαλία οι Εβραίοι, όταν τους έκαιγαν στην πυρά, τότε ε, βρήκαν ε, καταφύγιο στην Πολωνία. Στην ε, υπάρχει μια λέξη ε, και όπου η λέξη Πολωνία σημαίνει ότι μπορείτε να μείνετε εδώ. Και το 1948 όταν δημιουργήθηκε η χώρα του Ισραήλ, εγώ ήμουν ακόμη στο πανεπιστήμιο και θυμάμαι ότι είχα έναν Ισραηλινό φίλο, ο οποίο μου εξήγησε ότι οι Παλαιστίνοι έχουν αποκλειστικό δικαίωμα σε αυτή την ε, περιοχή, διότι ο Αβραάμ είχε τον αγαπημένο του ε, γιο. Και, και αυτή η διαμάχη από τη βίβλο εξακολουθεί να ισχύει και εδώ. Όταν ακούω λέξεις όπως το apartheid ή ακούω για παράδειγμα ότι το Ισραήλ διαπράττει εγκλήματα και βλέπω τα δεινά του Ισραηλινού εθνούς. Οπότε παρακαλώ μην ξεχνάτε πώς τους μεταχειρίστηκαν οι Παλαιστίνοι τρομοκράτες. Η Ευρώπη πιστεύει, πιστεύω χρειάζεται να κοιτάξει με έναν υγιή τρόπο την όλη κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Βόλας. Δεν τον βλέπω εδώ η κυρία Israel. Στο το Ισραήλ βρίσκεται σε μια πολύ ασταθή περιοχή στην Μέση Ανατολή. Εμείς τη λέμε να εγγύη Ανατολή στα γερμανικά, διότι είναι μόλι 3,5 ώρες πτήση από τη Βιέννη μέχρι το Τελαβίβ στην Ισραηλο-Παλαιστινιακή διαμάχη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ισραήλ περιβάλλεται από χώρε εχθρικέ που δεν θέλουν τίποτα άλλο παρά να το διαγράψουν από το τοπίο. Γι' αυτό το λόγο έχουν έναν από τους πιο σύγχρονους ε, ένα από τους πιο σύγχρονα συστήματα ασφαλείας ε, τον θόλο ασφαλείας γιατί πρέπει να υπερασπίσουν τη χώρα τους καθημερινά το Ισραήλ είναι η μόνη δημοκρατική χώρα στην περιοχή και αξίζει να έχει πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εταίρος μας και είναι η εγγύηση μας για ασφάλεια και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει ε, ω σημαντικό ε, συμμετέχοντα στην ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης και να θεωρείται ειλικρινή και ε, ισορροπημένο, ισόρροπο ε, Η κυρία Ward. Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν θεωρεί τους ε, Ισραηλινούς επικισμούς παρανόμους πλέον. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει ό,τι μπορεί για να αποσταθεροποιήσει και να θάψει τη λύση των δύο κρατών, βάζοντας την πρεσβεία της στην Ιερουσαλήμ και αναγνωρίζοντας την κυριαρχία του Ισραήλ στα υψίπεδα του Γκολάν. Οι επικισμοί είναι πάντα παράνομοι. Η έγκριση του Τραμπ δεν επηρεάζει το διεθνές δίκαιο και γι' αυτό ακριβώς είναι κάτι το οποίο υπονομεύει τις προοπτικές της λύσης των δύο κρατών και της αποκατάστασης της ειρήνης. Οι εκπρόσωποι των Παλαιστινίων πολύ σωστά καταδίκασαν την απόφαση αυτή σαν μια απειλή στην διεθνή τάξη και σαν την καταστροφή της λύσης των δύο κρατών. Πρέπει να έχουμε μια ενιαία θέση σε σχέση με τους επικισμούς, είναι παράνομοι, είναι εμπόδιο για την ειρήνη και υπονομεύουν τη λύση των δύο κρατών. Ζητάμε από την Ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει την εκτατική και αντιπαραγωγική της πολιτική στον τομέα των επικισμών. Ο κύριος Γόλας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Μογκερίνη, ασκήσατε κριτική στις παράνομες εγκαταστάσεις του Ισραήλ επανειλημμένα και καλά κάνατε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν πήρε μέτρα αποφασιστικά εις βάρος του Ισραήλ. Δεν ελέγχουμε εμείς ε, τα, τους τρόπους με τους οποίους οι Ηνωμένε Πολιτείες τους πείθουν να συμπεριφέρονται παράνομα εις βάρος των Παλαιστινίων και να προκαλούν γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Λέτε ότι υπάρχει ελπίδα για τη λύση των δύο κρατών. Πέθανε η λύση αυτή. Δεν σηκώνει πλέον ανάνυψης. Τώρα έχουμε μία λύση ενός κράτους μέσα στο οποίο και το Ισραήλ και η Παλαιστίνη θα πρέπει να έχουν ε, την δυνατότητα να χαίρουν μάλλον πλήρως των δικαιωμάτων τους και ταυτόχρονα να επιστρέψουν οι Παλαιστίνοι οι πρόσφυγες στα πατρικά τους εδάφη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε κάνουν αυτά που κάνουν μόνο και μόνο γιατί η Ευρώπη σε καμία περίπτωση δεν αντιδρά. Κύριε Τσουχουντάρο, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αυτή η φρικτή κατάσταση έχει διαρκέσει υπερβολικά, δυστυχώς. Αυτά που συμβαίνουν εκεί είναι απερίγραπτα. Εγώ είμαι γιατρός ε, στα επίγοντα και βλέπω ότι πέραν των πολιτικών παιχνιδιών χάνονται ζωές. Ε, είναι πολλά τα δεινά. Έχει έρθει η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο να φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όλους τους εμπλεκόμενους ούτω ώστε επιτέλου να βρεθεί μια δίκαιη λύση. Είχε περάσει υπερβολικά πολλή χρόνο. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει μια υγιή λύση, ούτω ώστε να σταματήσουν αυτά τα αποτρόπαια γεγονότα. Ελπίζουμε ότι αυτή η κατάσταση θα επιληθεί. Και η ελπίδα αυτή βρίσκεται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Αυτό ήταν ο τελευταίο ομιλητή για το Catch Δίνω τώρα το λόγο στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Υπετικπρόσωπο, για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλεια ε, την κυρία Μογκερίνη. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι σίγουρη ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο νέος ύπατος εκπρόσωπος θα σημειώσει και όλα όσα είπατε σήμερα εδώ σε αυτό το ημικύκλιο, αλλά να φροντίσει να διασφαλίσει και την ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των χωρών μελών. Να εμείνει στην ε, θέση μας όσον αφορά την προστασία του διεθνούς δικαίου, αλλά να συνεχίσει και τις σχέσεις και το συντονισμό και με άλλους στον κόσμο και το Ισραήλ αλλά και τον αραβικό κόσμο στην περιοχή. Ε, γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση και πιστεύω ότι με ρεαλισμό θα προχωρήσει. Είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρει να σκεφτεί και νέες πρωτοβουλίες προκειμένου να βοηθήσει να προχωρήσει η κατάσταση και να αποφύγουμε τα χειρότερα ε, που θα ήταν ε, χωρίς ε, τρόπο να κάνουμε πίσω. Σε μερικές περιπτώσεις και κάποιες στιγμές στην ιστορία απαιτείται οι δυνάμεις της ε, σοφίας να προσπαθούν να αποφύγουν τα χειρότερα και να μην έχουμε το φέα κομπλή, το πρωτετελεσμένο. Και οι καιροί που ζούμε τώρα ακριβώς απαιτούν από μας να παίξουμε αυτό το ρόλο. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να αποφύγουμε να πάνε τα πράγματα τόσο μακριά που οι θετικές προπτικές λύσεις της σύγκρουσης να μην υπάρχουν πια για το μέλλον. Ένα πράγμα θέλω να σχολιάσω που άκουσα στη συζήτηση και μου έκανε εντύπωση. Υπάρχει το θέμα των επικισμών αυτό καθεαυτόν, αλλά υπάρχει και το έργο μας, αυτό που κάνουμε και που θα συνεχίσουμε να κάνουμε, είμαι σίγουρη, ως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όσον αφορά την ε, σύγκρουση αυτή ε, Παλαιστίνης-Ισραήλ αλλά και αραβικού κόσμου Ισραήλ γιατί υπάρχουν δύο συγκρούσεις εδώ αλλά μην ξεχνάμε το ρόλο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύει και να προωθεί την τάξη που βασίζεται στο διεθνές Και κάποιος είπε εδώ ότι οι επικισμοί είναι αμφισβητούμενοι. Εγώ όμως έχω την εντύπωση ότι εδώ και ελπίζω τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην πηγαίνει προ αυτή την κατεύθυνση, όπου τελικά να αμφισβητούμε το ίδιο το διεθνέ δίκαιο. Αυτό θα ήταν πολύ επικίνδυνο. Οπότε δέχομαι ότι υπάρχουν διαφορές, αλλά πρέπει να ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να ε, βοηθήσουν απεμπλοκή στην, στην ε, περιοχή και τήρηση του διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο δεν είναι κάτι που συζητάμε, δεν αφισβητείται. Όταν φτάσουμε στη συζήτηση του κατά πόσο το διεθνές δίκαιο είναι καλό ή κακό, τότε ήδη έχετε πάει πάρα πολύ μακριά και έχετε φτάσει εκεί που δεν πρέπει να φτάνει ποτέ κανείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μαγκερίνη. Ολοκληρώνεται η συζήτηση για αυτό το θέμα. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση τη Αντιπροέδρου τη Επιτροπή, είπα τη εκπροσώπου τη Ένωση για θέματα εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, όσον αφορά την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένη τη κρίση στο Ιράν, το Ιράκ και το Λίβανο. Σα υπενθυμίζω ότι μπορεί κανεί να ζητήσει το λόγο στο Catch the Eye ή για μπλε κάρτα. Τι οδηγίε τι έχετε στην είσοδο του Μικυκλίου για μπλε κάρτα μόνο μετά, αφού έχουν μιλήσει δηλαδή οι πρώτοι ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Η συζήτηση αρχίζει με παρέμβαση της ε, Αντιπροέδρου και είπα της εκπρόσωπου εξωτερικής πολιτικής της κυρίας Μογκερίνη. μετά από επισκέψεις στη Βαγδάτη, στη Βηρητό και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής είδα ότι τα πράγματα εξελίσσονται. Ε, τα γεγονότα φαίνεται ότι και αυτά εξελίσσονται με γρήγορη ταχύτητα, οι διαμαρτυρίες πολλαπλασιάζονται ε, και έχουν σαν βασικό στόχο την ορθότερη διακυβέρνηση, την καταπολέμηση της διαφθοράς ε, και την οικονομική ευημερία. Εμείς καταδικάζουμε όλες τις πράξεις βίας από οποιαδήποτε πλευρά και αν προέρχονται, ζητάμε τον σεβασμό της ελευθερίας έκφρασης και την άμεση διερεύνηση των αιτιών της, των φαινομένων βίας. Τώρα να κάνω κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις ε, σχετικά με αυτά τα οποία ήδη ακούστηκαν και για το Ιράκ. Το Ιράκ αντιμετωπίζει πολύ ειδικά προβλήματα. Έχει ανάγκη από αποκατάσταση της ειρήνης, έχει ανάγκη από ανοικοδόμηση, έτσι ώστε να υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες για όλους. Αυτά είναι απαραίτητα εάν το Ιράκ σταθεροποιηθεί μακροπρόθεσμα και έχουν μένει πολλά να γίνουν και στον τομέα της συμφιλίωσης και της ανοικοδόμησης. Από την άλλη βήματα προόδου έχουν ήδη σημειωθεί. Εμείς από την αρχή των προβλημάτων ζητήσαμε διάλογο ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, όπως πρότεινε άλλωστε και η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να ζητήσουμε την κυβέρνηση του Ιράκ να συνεχίσει την προσπάθεια επικοδομητικής συνεργασίας με όλες τις χώρες της περιοχής. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις χώρες του Ιράκ να κερδίσουν την ειρήνη, θα συνεχίσουμε να το στηρίζουμε έτσι ώστε να οδηγηθούν σε μια δημοκρατία χωρίς αποκλεισμούς. Για το Ιράν τώρα υπάρχουν και εκεί διαδηλώσεις λόγω της παρούσης οικονομικής δυσκολίας. Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα ειρηνικής διαδήλωσης και δεν είναι σε καμία περίπτωση δικαιολογημένη υπερβολική βία των αρχών. Θα πρέπει να υπάρξει άμεση διερεύνηση των αιτιών της βίας αυτής έτσι ώστε να υπάρξει ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών και πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς διακοπές. Να προσθέσω κάτι που είναι προφανές, ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την εφαρμογή μη της Συμφωνίας για τον πυρο...